Καλησπέρα σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμότατα όλους και ελπίζω η θερινή αυτή ανάπαυλα να σας ε, γέμισε τις μπαταρίες και να γυρίσετε ακμεότατοι για το τελευταίο σημαντικό αυτό τρίμηνο του χρόνου γιατί κατά τη διάρκεια του θα ολοκληρώσουμε και τους εκρεμείς τριμερείς διαλόγους για τη συνοχή. Για τη σημερινή μας συνεδρίαση, θα σας πρότεινα δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε με το σημείο 9 της σημερινής διάταξης, προκειμένου να προλάβουν οι συνεισηγητές να μας παρουσιάσουν το έγγραφο εργασίας τους. Γιατί η Κωνσταντ Κρέλ, μία από τις συνεισηγητές, έχει άλλη συνεδρίαση μετά. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξή μας με αυτή την αλλαγή που σας πρότεινα. Επίσης, θα ήθελα να σας ζητήσω να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 6ης Ιουλίου του 2020. Ε, υπάρχουν στο διαδίκτυο. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα σας πρότεινα ο συνήθως να θεωρήσουμε ε, ως συγκεκριμένα τα πρακτικά. Και να περάσουμε αμέσως, όπως σας πρότεινα, στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, που αφορά το κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Ξέρετε πόσο σημαντική είναι αυτή η νομοθετική πράξη για την, και για τη δική μας Επιτροπή. Και ε, ο νέος κανονισμός για το 2021-2027 παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2018 και μετά από πολλοί μήνες εργασίες και στην Επιτροπή μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το Μάρτιο του 2009 την θέση του για την πρώτη ανάγνωση. Τη θέση που αποτελεί και τη διαπραγματευτική μας εντολή. Και τον Ιανουάριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει την νομοθετική της πρόταση για να περιλάβει και το νέο Ταμείο Δικής Μετάβασης στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Στη συνέχεια, το Μάιο και μετά από έτοιμα της δικής μας Επιτροπής και στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, προτείναμε να ληφθούν κάποια κατεπήγοντα μέτρα οι συγητές ε, του κανονισμού περί κοινών διατάξεων προτείνουν ένα έγγραφο εργασία με τη θέση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των νέων ε, αλλαγών του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, όπως είχαμε αποφασίσει στη συνεδρίαση των συντονιστών και στην Ολομέλεια της Επιτροπής μας. Υιοθετήσαμε μετά από συζήτηση στη διαπραγματευτική μας ομάδα με συμφωνία των σχεδόν εισηγητών των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Θα δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο, αν το επιθυμούν φυσικά, στους συνεισηγητές μας για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων για να μας κάνουν την παρουσίαση του εγγράφου της. Ο ένα από τους δύο συνεισηγητές είναι ο Αντρέι Νοβάκοφ. Θα μιλήσει πρώτα αυτός και κατόπιν η Κωνσταντζε Κρέλ για να μας κάνει και εκείνη τα σχόλιά της. Πρώτα λοιπόν θα ακούσουμε τον Αντρέι Ναβάκοφ, που δεν έχει έρθει όμως από ό,τι βλέπω, οπότε ας ακούσουμε πρώτα την κυρία Κωνσταντσε Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, κρίμα ε, που ακόμα συναντώμαστε ε, στο πλαίσιο του remote. ελπίζω ότι μετά το ε, διάλειμμα του καλοκαιριού θα ηρεμούσε η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά λειτουργεί. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είχαμε μια συζήτηση σχετικά με την ολοκλη... στο CPR το... τα θέματα τα οποία αφορούν το πεδίο εφαρμογής για τον κανονισμό πυρκινών διατάξεων ε, ε, ε, υιοθετήσαμε τις προτάσεις, της τροπολογίας της Επιτροπής, συζητήσαμε με τον εισηγητή, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διαφωνίες. Επίσης, καταστήσαμε εφικτό ότι θα υπάρξει ένας διορθωτικός ε, διάλογος ε, μαζί με την Επιτροπή σε περίπτωση που υπάρξει έκτατη ανάγκη για κάτι τέτοιο, όμως αυτό θα γίνει μονάχα σε κατάσταση ε, που είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι ε, να ε, συμπεριλάβουμε το συγκεκριμένο έγγραφο ε, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και στην συνέχεια να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την τρομερή διάλεγη. Αυτά από πλευρά μου. Ελπίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή θα το λάβει υπόψη της ε, ε, το έγγραφο αυτό ακριβώς όπως έκαναν και οι σκιώδεις. Ευχαριστώ πολύ σε αυτό το σημείο επίσης για την πολύ καλή εργασία από πλευράς ε, των πολιτικών συμβούλων, των βοηθών της γραμματείας όσον αφορά του React-EU. Έτσι μπορούμε σήμερα να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή για το θέμα αυτό και το ότι είναι εφικτό το να... Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, μπορούμε να ψηφίζουμε σήμερα σε αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους μας βοήθησαν. Ήταν ε, κάτι το ασυνήθιστο εν μέσω των καλοκαιρινών ε, διακοπών και όλα έγιναν ε, ουσιαστικά με μία συνάντηση των σχεδόν ε, και στη συνέχεια γινόταν ε, γραπτές ανταλλαγές μηνυμάτων όπου δηλώνουμε τις θέσεις μας σχετικά με το προσχέδιο για το ReactEU και θα χαρώ πολύ αν η ψηφοφορία θα είναι και θετική σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Merci Σας ευχαριστώ, αγαπητή Κωνσταντζε Κρέλ και ευχαριστώ και εκ μέρους του προσωπικού για τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες και ευχαριστώ και εγώ θερμά και εσένα για το πολύ αξιόλογο έργο σου και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Κυρίως για το React EU που θα εξετάσουμε αργότερα. Θέλει παρακαλώ άλλος κάνει το λόγο? Δεν βλέπω κανένα συνάδελφο να θέλει το λόγο. Δεν έχει εμφανιστεί και ο Αντρέι Νοβάκοφ, οπότε θεωρούμε ότι λίγη συζήτηση για το θέμα αυτό και θα περάσουμε στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως. Και μια και πρόκειται για ενδεικτική ψηφοφορία, ε, για να δώσουμε την πολιτική μας έγκριση για το έγγραφο, θα γίνει μια ενιαία ψηφοφορία για το σύνολο του εγγράφου. Και η ψηφοφορία εξ αποστάσεως θα γίνει με το σύστημα iVote. Τα αποτελέσματα θα σας ανακοινωθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 2 παρατέταρτο και θα ολοκληρωθεί στις 3 παρατέταρτο. Ενώ η τελική ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 3 και 4 και θα ολοκληρωθεί στις 4 και 4. Και επαναρχόμαστε στην κανονική σειρά των σημείων της ημερήσιας διάταξης με το σημείο 4 την πρόταση απόφαση του Συμβουλίου που επιτρέπει στη Γαλλία να εφαρμόσει για κάποιους έμεσους φόρους ένα μειωμένο συντελεστή φορολογικό στο παραδοσιακό ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάννα, τη Μαρτινίκα και τη Ρενιό. Οι προτάσει αυτέ αφορούν το επόμενο πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο του 2021 με 2027. Και όπω ξέρετε, στηρίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτρέπει κάποιες παρεκκλήσεις ε, ε, από τις ε, συνθήκες και τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα υπερπόντια διαμερίσματα προκειμένου να αντισταθμιστούν κάποια φυσικά τους μειονεκτήματα και ιδιαίτερες δυσκολίες που έχουν. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά το ρούμι που παράγεται στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα. Και μάλιστα το κείμενο αυτό δεν είναι καινούριο ή πρωτοφανέ. Παρόμοιε παρεκκλήσει ε, εφαρμόζονται με τον ΑΒ τρόπο από το 1923 και αντισταθμίζουν εν μέρη το υψηλότερο κόστος παραγωγής στα υπερπόντια διαμερίσματα. Και η προτινόμενη απόφαση θα επιτρέψει τη Γαλλία να μειώσει του ειδικού φόρου κατανάλωση και τι εισφορέ τη κοινωνική ασφάλισης για το παραδοσιακό ρόμι που παράγεται στη Γοδελούπη, τη Γαλλική Γουιάννα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιό και πολίτε στι περιοχέ αυτέ ή στη Μητροπολιτική Γαλλία. Και οι μειώσει αυτέ θα αφορούν το πολύ 50% του κανονικού συντελεστή. Η προτινόμενη παρέκκληση δικαιολογείται γιατί το πεδίο εφαρμογή τη είναι εξαιρετικά περιορισμένο και επίση δικαιολογείται από τι οικονομικέ δυσκολίε που είναι εγγενεί ε, τη παραγωγή στα υπερπόντια αυτά διαμερίσματα που σα ανέφερα. Και άλλωστε η παρέκκληση αυτή συνάδει πλήρω με την ανάλυση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τις ε, αρχές του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υποφαινόμενος ως εισηγητής και μετά από διαβουλεύσεις με τους συντονιστές θα πρότεινα, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν για τέτοιου του θέματα, ε, ο κανονισμός ε, να εξεταστεί δυνάμει το άρθρο 52, παράγραφος 1 του κανονισμού, με την απλοποιημένη δηλαδή διαδικασία η έγκριση του κανονισμού να γίνει με την απλοποιημένη διαδικασία χωρίς τροπολογίες. Μάλιστα το σχέδιο έκθεσης σας έχει ήδη μοιραστεί και πριν περάσουμε στην έγκριση της διαδικασίας αυτής θα ήθελα να ρωτήσω αν θα ήθελε κάποιος συνάδελφος το λόγο. Όχι. Στην αίθουσα τουλάχιστον. Κάποιος εξ αποστάσεως θα ήθελε το λόγο μήπως. Όχι. Οπότε σας ζητώ και επίσημα να μου πείτε αν έχετε αντιρρήσεις ως προς την υιοθέτηση του κανονισμού αυτού με την απλοποιημένη διαδικασία. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Και μια και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την απλοποιημένη διαδικασία, εγκρίνουμε την έκθεσή μου με τη διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ θερμά και περνούμε αμέσως στο επόμενο σημείο, το σημείο 5 τη δεύτερη απόφαση που αφορά το φόρο IEM για την αγορά και διάθεση προϊόντων στις Κανάριες νήσους. Πρόκειται για μερική ιολική ε, απαλλαγή από το φόρο για κάποια τοπικά προϊόντα, μια παρέκκληση που ισχύει από το 2002 και που αντισταθμίζει μερικώς το υψηλότερο κόστος παραγωγής λόγω της απομόνωσης, ε, της μεγάλης απόστασης ε, των Κανάριων νησιών από τη Μητροπολιτική Ισπανία. Και οι απαλλαγές αυτές ε, δεν μπορούν να επηρεάζουν την τιμή των προϊόντων το πάνω από 15% ούτε να ξεπερνάνε ένα ετήσιο ανώτατο όρο 150 εκατομμύριων ευρώ. Αυτές οι φορολογικές εξαιρέσει και παρεκκλήσει, δικαιολογούνται από το πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογή του και από τις ε, εγγενείς οικονομικές ε, δυσκολίες ε, των της παραγωγής των Καναρίων Ίσων. Άλλωστε, οι παρεκκλήσεις αυτές συνάδουν πλήρως με την ανάλυση που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εισηγητής για το θέμα αυτό, και μετά από διαβούλευση με τους ε, συντονιστές θα ήθελα και πάλι να σας προτείνω να εγκρίνουμε τον κανονισμό αυτό με την απλοποιημένη διαδικασία δυνάμει του άρθρου 52 παράγραφος 1 και μάλιστα χωρίς τροπολογίες. Το σχέδιο έκθεσης σας έχει ήδη μοιραστεί και θα ήθελα να ρωτήσω αν θα ήθελε κανείς το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω, ούτε στην αίθουσα ούτε εξ αποστάσεως. Οπότε, ερωτώ και επισήμως, υπάρχουν αντιρρήσεις ε, στην έγκριση του κανονισμού αυτού με την απλοποιημένη διαδικασία. Όχι, ούτε στην αίθουσα, ούτε εξ αποστάσεως. Και μια και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε την έκθεση. Και σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα σε μια άλλη έκθεση. Είναι το μεσημέρι των ε, υπερπόντιων περιοχών και των εξόχως κέντρων περιοχών. Ε, περνάμε λοιπόν σε άλλο ένα σχέδιο έκθεσης που αφορά τα υπερπόντια γαλλικά εδάφη και αφορά την εισφορά θαλάσσης. Είναι ένας φόρος που εφαρμόζεται σε πωλήσει στα υπερπόντια γαλλικά εδάφη. Η εξαίρεση αυτή που γνωρίζουμε πολύ καλά στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης επιτρέπει μειωμένους φόρους για ορισμένα προϊόντα που παράγονται τοπικά ούτω ώστε να αντισταθμίσουν το οικονομικό ε, μειονέκτημα και να ενισχύσουν την τοπική παραγωγή. Οι γαλλικές αρχές έχουν ζητήσει ανανέωση της ε, απαλλαγής για την περίοδο 2021-2027. Ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες αξιολογήσεις ούτε όλες οι μελέτες ε, που επιβάλλονται λόγω της επιδημίας COVID-19. Η Κομισιόν λοιπόν προτείνει το σημερινό καθεστώς το οποίο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2021 να παραταθεί κατά ένα εξάμεινο, ούτως ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος για τις γαλλικές αρχές να μπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτή την έκθεση που είναι πολύ σημαντικά και μετά το θα γίνει εκ νέου διαβούλευση με το Κοινοβούλιο για το καθεστώ αυτό του χρόνου, το επόμενο το συγγνώμη. Αυτή η εξαίρεση, αυτή η απαλλαγή ε, σε σχέση με τους φορολογικούς κανόνες ε, δικαιολογείται χάρη στο περιορισμένο, τρομακτικά περιορισμένο πεδίο εφαρμογή και συμμορφώνεται απόλυτα με το άρθρο 349 της συνθήκης. Ως συνεισηγητής και μετά από διαβούλευση με τους συντονιστές θα προτείνω εκ νέου να εφαρμοστεί το άρθρο 52.1 για τον κανονισμό αυτό, δηλαδή η απλοποιημένη διαδικασία χωρίς τροπολογίες. Το σχέδιο έκθεση σας έχει διανεμηθεί. Θα ήθελε κάποιος συνάδελφος να εκφράσει κάποια άποψη εδώ στην αίθουσα ή από απόσταση. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Θα σας ζητήσω λοιπόν επισήμως αν υπάρχουν ενστάσεις ε, για την υιοθέτηση αυτού του κανονισμού με την απλοποιημένη διαδικασία. Υπάρχουν ενστάσεις, όχι, δεν βλέπουμε να υπάρχουν ενστάσεις. Η έκθεση συνεπώς εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία με τη διαδικασία εξαποστάσεως ψηφοφορίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι κανόνες παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς ε, που εφαρμόστηκαν και πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Σήμερα στην Επιτροπή Ρέτζι έχουμε τρεις ε, ψηφοφορίες. Μία πάρα πολύ σημαντική αφορά το React.eu και δύο άλλες ψηφοφορίες που είναι εξίσου σημαντικές ε, για την νέα μηχανική στρατηγική και για τον ε, κανονισμό των γενικών διατάξεων. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στις ψηφοφορίες βάσει δύο βήματων. Πρώτα οι τροπολογίες για τα δύο πρώτα θέματα, Reactive και νέα βιομηχανική στρατηγική. Και σε δεύτερη φάση θα έχουμε την τελική ψηφοφορία και για τα τρία θέματα. Η ψηφοφορία για τις τροπολογίες είναι ανοιχτή έω τι 3 παρατέταρτο, 2 και 45. Η γραμματεία στη συνέχεια θα μα ενημερώσει μέσω mail ποιε τροπολογίε έχουν εγκριθεί και ποιε έχουν απορριφθεί. Στη συνέχεια θα λάβει χώρα η τελική ψηφοφορία από τι 3 και 4 έω τι 4 και 4. Μετά από την τελική ψηφοφορία, η γραμματεία θα μα ενημερώσει ξανά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία. Για κάθε ψηφοφορία και το συγγνώμη που το επενθυμίζω πρέπει ο καθένας σας ξεχωριστά να ψηφίσει στην εφαρμογή iVote προσωπικά και να στείλει το υπογεγραμμένο ψηφοδέλτιο στη γραμματεία. Μόνο οι μόνιμοι ε, ευρωβουλευτές ε, και οι αναπληρωτές που έχουν οριστεί πριν από την ε, προθεσμία που ορίστηκε την περασμένη Παρασκευή στην κάθε πολιτική ομάδα μπορούν να ψηφίσουν. Τρία τελευταία σημεία, πολύ σημαντικά πριν ξεκινήσετε την ψηφοφορία. Κάθε ευρωβουλευτής μπορεί να ψηφίσει μόνο μία φορά. Δεν μπορείτε να ξαναψηφίσετε στο iVote εκτός αν έχετε κάνει κάποιο λάθος στην πρώτη ψηφοφορία. Δεύτερον, κάθε ευρωβουλευτής πρέπει υποχρεωτικά να στείλει και το ψηφοδέλτιό του σε υπογεγραμμένο αρχείο μορφής PDF από το προσωπικό του email του Ευρωβουλευτή, δηλαδή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη Γραμματεία και αυτό πριν κλείσει η ψηφοφορία στι 14.45. Διαφορετικά η ψηφοφορία δεν είναι ούτε επαληθεύσιμη ούτε έγκυρη. Η ψήφο, συγγνώμη. Και εκεί μπορεί. Τέλο, για να ταυτοποιηθεί η ψηφοφορία χρειάζεται ο αριθμητικό κωδικό που βρίσκεται πάνω δεξιά στο ψηφοδέλτιο. είναι προτιμότερο να υπάρχει μία υπογραφή επί της οθόνης παρά ε, με σκαναρισμένη. Οι άλλες ε, πληροφορίες ε, σας έχουν σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη γραμματεία. Δεν θα τις επαναλάβω λοιπόν. Είναι αρκετά περίπλοκα έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Τα γνωρίζετε όλα. Οπότε τώρα πάμε στην συνοπτική παρουσίαση των κειμένων και των ψηφοφοριών. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, το πολύ σημαντικό σημείο που εξετάζει η Επιτροπή μας ε, σήμερα το μεσημέρι, αφορά το react και δίχως άλλο πρόκειται για ένα από τα πλέον επίγοντα θέματα αυτή την εποχή στην Επιτροπή μας. Αφορά τη διάθεση 55 δισεκατομμύριων ευρώ για την ανάκαμψη μετά την επιδημία συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού έτους που τρέχει αυτή τη στιγμή. Ε, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ε, ε, επιταχυμένη για αυτό το φάκελο. Μας υπέβαλαν το σχέδιο έκθεσης συνεισηγητές τον Ιούλιο. Οι τροπολογίες μεταφράστηκαν κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Οι συμβιβασμοί, οι συμβιβαστικέ που επιτεύχθηκαν επιτεύχθησαν πάρα πολύ γρήγορα με τη συμμετοχή όλων και όπως είπε η Κωνσταντ Κρέιλ προηγουμένως θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλη τη γραμματεία για τις ε, προσπάθειες που κατέβαλε αλλά κυρίως θα ήθελα να συγχαρώ τους ε, εισηγητές των Αντρέι Νοβακόφ και την Κωνσταντσε Κρέιλ για τις άριστες προσπαθίες τους και το άριστο αποτέλεσμα κατά τις διαπραγματεύσεις ε, που θα λάβουν χώρα πολύ σύντομα όπως θα σας πω σήμερα το μεσημέρι, θα έχουμε κάποιο θέμα που θα μας απασχολήσει. Αρκετά σημαντικό. Διότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν μεταξύ τους για να μην γίνουν τροπολογίες στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Κάτι που εκ των πραγμάτων περικόπτει τα 5 πρώτα δισεκατομμύρια για το 2020 από το ReactEU. Όπως φαίνεται το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο στην παρούσα φάση να αλλάξει άποψη. Γνωρίζουμε λοιπόν ε, στο εξή ε, ότι οι τρίλογοι πρόκειται να ξεκινήσουν και να ασχοληθούν με αυτό το πρόβλημα. Και μπορώ να σας πω με σχετική βεβαιότητα ότι το Κοινοβούλιο δεν θα δεχθεί αυτές οι διατάξεις που αντιτίθεται με, αντίκειται στα συμπέρασματα του Συμβουλίου θα καταφέρουν ε, να δοθούν 2,5 δισεκατομμύρια ή παραπάνω στο ReactEU. Εμείς ε, έχουμε στείλει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμών ε, και στους πρόεδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να τους ενημερώσουμε για το πρόβλημα αυτό το οποίο είναι πολιτικού χαρακτήρα αλλά και δημοσιονομικού. Δίνω αυτή τη στιγμή το λόγο λοιπόν στους συνεισηγητές. Πρώτα απ' όλα στην Κωνσταντ Κρέλ, η οποία εξακολουθεί να είναι μαζί μας και σας ευχαριστώ. Κωνσταντ Κρέλ, έχετε το λόγο. Από ό,τι βλέπω η Κωνσταντ Κρέλ είναι συνδεδεμένη αλλά με είχε ενημερώσει ότι είχε κάποια άλλη συνεδρίαση και ότι ίσως θα δυσκολευόταν να είναι παρούσα σε αυτή τη συζήτηση για το Reactive οπότε δίνω το λόγο στο συνεισηγητή μας, αν είναι μεταξύ μας, ε, ανάμεσά μας, τον Αντρέι Νοβακόφ. Bon. Andrei. Ναι. Ούτε ο Ανδρέη βρίσκεται εδώ. Έχουμε ήδη κάνει κάποιες συζητήσεις για το θέμα αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για την ψηφοφορία σήμερα, οπότε ε, ξεκινάει η διαδικασία ψηφοφορίας και πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης που αφορά τις νέες βιομηχανικές στρατηγικές για την Ευρώπη. Η Κομισιόν επίση ε, θα ψηφίσει σήμερα τη γνωμοδότησή τη ε, όσον αφορά την έκθεση πρωτοβουλία τη ΙΤΡΕ για μια νέα στρατηγική μακροχρόνια για το βιομηχανικό μέλλον τη Ευρώπη. Η εισηγήτριά μα, η συνάδελφο κυρία Πένκοβα, ασχολήθηκε με το θέμα. 125 τροπολογίε ε, υποβλήθηκαν έγκαιρα και η εισηγήτρια και ο σκιώδη εισηγητή συμφώνησαν για τρει συμβιβαστικέ τροπολογίε ε, τροπολογίε. τροπολογίες. Η κυρία Πάνκοβα θα ήθελε να πάρει το λόγο ε, πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Ζητάει κάποιο το λόγο, ζητάει η κυρία Πάνκοβα το λόγο. Όχι, όπως φαίνεται. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία για την έκθεση αυτή, αφού η διαδικασία ψηφοφορίας έχει ανοίξει. Υπάρχουν ερωτήσεις ε, για τα διάφορα από τα μέλη. Όχι, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Πολύ ωραία. Ήμασταν λοιπόν ταχύτατοι, πολύ περισσότερο γρήγοροι από ό,τι θα είχα φανταστεί. Μια χαρά οργανωμένοι είμαστε. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020 από τις 13 και 45 έως τις 15 και και ότι αυτή τη συνεδρίαση θα ακολουθήσει μια συνεδρίαση συντονιστών όπου θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις ως επιτοπλίστων ε, για την ανάκαμψη, τη συνέχιση και τη, μάλλον των διαπραγματεύσεων που έχουν ξεκινήσει με το Συμβούλιο. Και θα γίνουν και κάποιες ανταλλαγές απόψεων μετά από το τελευταίο, ε, επί του τελευταίου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και θα ζητήσω από τους συντονιστές ε, να έχουν την καλοσύνη να βρίσκονται εδώ στις 2.45 ε, για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ όλους.